Καλημέρα σας. Ελπίζω από την κυρία Χαϊόνι Βίστ να μπορεί να περάσουν στο δεύτερο τμήμα επειδή δεν έχουν φτάσει οι ενδιαφερόμενοι για το πρώτο. Τώρα, πρώτα απ' όλα, ανακοινώσει τη Προέδρου. Χθε λάβαμε μια επιστολή του κυρίου Σούλτσου. που μα ενημέρωσε για την απόφαση του διάσκεψη των Προέδρων της 12 Δεκεμβρίου για ενδεχόμενη συμβολή του Λίμπερ Σνόουντεν στην ε, Επιτροπή Λίμπε. Εστάλει λοιπόν ένα κοινωνικό ταχυδρομείο σε όλα τα κράτη, σε όλες, συγνώμη, σε όλες τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής μας. Και Εάν η Επιτροπή μας λάβει απόφαση να ε, δεχθεί τις εργασίες του Σνόντον, θα το δεχθούμε, διαφορετικά εάν υπάρξουν προβλήματα θα δεχθούμε μια μαγνητοφωνημένη, μαγνητοσκοπημένη παρουσίαση. και οι συντονιστές ε, θα κληθούν σήμερα να αναφέρουν την θέση τους ε, μέσω γραπτής διαδικασίας. Αυτή ήταν η ανακοίνωση λοιπόν που είχα να σας πω. Αλλάζουμε τα σημεία στη μέσα διάταξη, θα ξεκινήσουμε με την έκθεση κυρίας Βαϊόν. τρίτε χώρε οποίων οι υπήκοοι υπόκειται σε υποχρέωση θεώρηση για τη διέλευση εξωτερικών συνόρων και τρίτε χώρε οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή. Θα ακούσουμε την πρόταση από την Κομισιόν και μετά η κυρία Φαγιών θα λάβει το λόγο και μετά η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα. Νομίζω ότι μπορεί να είμαι ιδιαίτερα σύντομο, διότι αυτή η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει την μετακίνηση των επικών ε, αυτής της χώρας ε, στο πλαίσιο της ε, συμφωνίας που έχει υπογραφεί το 2010 πρόκειται για ένα διάλογο ο οποίος αφορά την απελευθέρωση από τη θεώρηση όπως ξέρετε αφορά τέσσερα μπλοκ αυτό σημαίνει πως ε, ένα πρώτο μπλοκ αφορά τα βιομετρικά στοιχεία το δεύτερο μπλοκ για την ε, παράτυπη μετανάστευση συμπεριλαμβανομένως της το ε, τρίτο μπλοκ για την δημόσια ασφάλεια και την δημόσια τάξη και ασφάλεια αυτή η μεθοδολογία η Κομισιόν πάνω την ακολούθησε σε όλες τις ε, διαλόγους για την κατάργηση των ε, προξενικών θεωρήσεων και περίπτωση αυτή της ε, Μολδαβίας πρόκειται για τις σχετικές απαιτήσεις που βλέπουν εκθέσεις, υποβολή εκθέσεων, των οποίων πέντε έχουν ήδη εγκριθεί, έχουν γίνει κάποιες αποστολές των δημοκρατία της Μολδαβίας όπου θέσαμε κάποια ορόσημα ειδικά στο πλαίσιο του δεύτερης φάσης του πρόγραμματος δράσης το ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Μολδαβοί αν θέλουν να έχουν αυτήν την ε, θεώρηση δωρεάν συζήτηση διεξάγεται και στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο που αφορά την πρόταση της Κομισιόν για την μεταφορά στην ε, κατάλογο των θεωρήσεων ε, δωρεάν, της παρέχης δωρεάν ε, θεωρήσεων και η πρόταση αυτή βρίσκεται υπό συζήτηση και σύντομα θα έχουμε τριμερείς διαλόγους. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στο αφορά την απελευθέρωση του θεωρήσεων για τη Μολδαβία και του διαλόγου που διεξάγεται και την 13 Νοεμβρίου η πέμπτη έκθεση ολοκληρώθηκε η Κομισιόν ανέφερε ότι πληρούνται όλες τις προϋποθέσεις από τη Μολδαβία σε αυτή τη φάση. Γι' αυτό λοιπόν υποβάλλουμε αυτή την πρόταση που προβλέπει την μεταφορά των πολιτών στην διαδικασία της ελεύθερης θεώρησης, αλλά αυτό θα εφαρμόζεται σε όλους τους πικούς που διαθέτουν βιομετρικά στη ε, διαβατήρια. Ε, στο της κορυφής του Βίλνιους ε, συζητήθηκε το θέμα διότι η Επιτροπή θέλει να, θέλει να δώσει ένα πολιτικό μήνυμα ότι η Κομισιόν ε, τιμά τις υποχρεώσεις της ε, και γι' αυτό υποβάλαμε την πρόταση να μετακινηθεί η χώρα αυτή στην ε, κατάλογο των χωρών που έχουν τις ελεύθερες, που διαθέτουν ελεύθερη θεώρηση. Το, το, το, Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβουν τις ευθύνες τους. Εμεί θα ήμασταν υπέρ μιας ε, έγκρισης ε, της πρότασης για να δείξουμε στη Μολδαβία πως ε, επαναλαμβάνω η Ευρωπαϊκή Ένωση τιμάει τις υποχρεώσεις της και να ολοκληρωθεί ο φάκελος αυτός κατά τη διάρκεια της θητείας ε, του Κοινοβουλίου πριν δηλαδή ολοκληρωθεί. Θα διεξαχθεί και άλλη μια συνεδρίαση του Συμβουλίου ΔΕΗ και τα πράγματα βαίνουν καλώς προς το παρόν και ελπίζουμε πως το Συμβούλιο θα μπορέσει να δεχθεί την πρόταση. Ένα τελικό σημείο. Πολλά ελέγχθησαν σχετικά με την κατάκριση αυτού του συστήματος του Visa Free μετά από την διαδικασία απελευθέρωσης ε, του θέματος της χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα, στις αρχές Ιανουαρίου, θα τεθεί σε εφαρμογή ο μηχανισμός ε, περί θεωρήσεων και αυτή η απελευθέρωση θα μπορεί προσωρινά να ανασταλεί. Παναλαμβάνω ότι απαιτούν, απαιτείται διάθεση βιομετρικών διαβατηρίων και κατά άποψη της Κομισιόν θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε επί του ζητήματος αυτά. Με ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην κυρία Βαϊόντ, συγγήτρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτής της έκθεσης και για την ενημέρωση για τα όσα τεκτενώνει στο Συμβούλιο. Ήμουν εισηγήτρια για το θέμα της θεώρησης των πολιτών της Μολδαβίας μετά από τα όσα συνέβησαν με τις, αυτά με τα γεγονότα με τις χώρες της Δυτικών Βαλκανίων όπως είπατε είναι πολύ σημαντικό να στείλουμε ένα θετικό και ισχυρό πολιτικό μήνυμα στον Μολδαβία ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του διάσκεψης κορυφής του Βίλνιους σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον και η δημοκρατία της Μολδαβίας ε, ετοιμάστηκε εδώ και τρία χρόνια για την ε, υποδοχή αυτής της διαδικασίας ε, και χαίρομαι που αναφέρει η Κομισιόν ότι όλες τις προϋποθέσεις η ελεύθερη διακίνηση είναι ένα θεμελιώδες ε, ευρωπαϊκό δικαίωμα και γνωρίζοντας την ε, εμπειρία του παρελθόντος στην χώρα αυτή και γενικά στις νέες χώρες που έχουν ταχθεί στο σύστημα για να είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ολοκληρώσουμε διαδικασία στι αρχέ ε, τη Άνοιξη ε, και πριν από τη λήξη τη θητεία του Κοινοβουλίου. Περιμένω λοιπόν μια πολύ καλή συνεργασία με τους πιο εισηγητέ αλλά και με το Συμβούλιο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειε τώρα του ζητήματο ότι θα έχουμε την παρουσίαση της εκθέσεως στι 19 ε, Ιανουαρίου και αν όλα πάνε καλά ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Φεβρουάριο θα ήθελα να πω ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το καθεστώς των θεωρήσεων διότι είναι πολύ σημαντικό να στηρίξουμε την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Πρόθεσή μου είναι να ολοκληρωθεί ο φάκελος συντομό δυνατών με την ελπίδα πως ε, η Μολδαβία θα πληρεί όλα τα απαραίτητα κριτήρια τώρα για την ε, ρήτρα προφύλαξης, ε, για μηχανισμό ε, ανα, ανάκλησης. Ελπίζω ποτέ να μην βρεθούμε στη θέση να τον χρησιμοποιήσουμε. Ειδικά διότι όταν μιλάμε για κράτη των Δυτικών Βαλκανίων θα ήταν ένα πολύ, πολύ σημαντική επιστοδρόμηση εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός ακόμα και αν πρόκειται για προσωρινή ανάκληση. Διότι αν δείτε αφετέρου το θέμα των ετούντων άσυλο τον οποίο ο αριθμό ε, δεν είναι μειούμενο συνεχώ, νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φαγιόν. Το ζήτημα της κατάχρησης των θεωρήσεων, των εξαίρεσης θεωρήσεων, μπορεί να μην προβλέπεται. Αν βλέπουμε όμως τα κράτη ε, τα, σύμφωνα με το κεφαλήν εισόδημα στις ε, χώρες αυτές θα ε, λέγαμε ότι αυτή η κατάχρηση είναι μάλλον προβλέψιμη. Ή γίνει καμιά μελέτη αναφορικά με την ε, κατάχρηση αυτού του καθεστώτος ε, ελεύθερων θεωρήσεων. Εάν δεν υπάρχουν θεωρήσεις, τότε θα είναι δυνατόν να επιδεινωθεί η υπόθεση. Ευχαριστώ κύριε Βέμπερ. Ευχαριστώ πρόεδρε να καλωσορίσω αυτή την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφραστεί για ένα παρόμοιο καθεστώς θεωρήσεων με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και είμαι πεπισμένη πως ε, αυτό θα οδηγήσει σε μια ενισχυμένη συνεργασία εντός εισαγωγικών ανάμεσα στην κυβέρνηση της Μολδαβίας και την ε, Κομισιόν διότι κρίνω πως ε, είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε όχι μόνο τον κύριο Μπρόγκ αλλά και άλλους οι οποίοι ανησυχούν ότι θα συμβεί η αποκάλυψη στην, ε, στην Ευρώπη νομίζω πως το θέμα θα πρέπει να ειδωθεί στο σύνολό του και είναι όντως η νέα διαδικασία ή μάλλον η ανάκληση θα τον ε, θεωρήσουν, θα τεθεί σε ισχύ, θα υπάρχει δυνατότητα λοιπόν και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Κομισιόν και την ε, κυβέρνηση ιασδήποτε τρίτης χώρα με αυτό το καθεστώς ε, ελεύθερης θεώρησης. Να πω επίσης πως όσοι θέλουν να εγκαταλείψουν τη χώρα προέλευσης, τη χώρα καταγωγής τους, το έχουν ήδη πράξει. Τώρα μιλάμε για τον υπόλοιπο πληθυσμό, επιπλέον το, να διαθέτει κάποιος βιομετρικό διαβατήριο, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσει την όλη διαδικασία από την αρχή, κάτι το οποίο δεν είναι πολύ απλό και εύκολο. Γι' αυτό λοιπόν είμαι πολύ πεπισμένοι πως αυτό θα πρέπει να αποβαίνει προς όφελος των πολιτών της Μολδαβίας και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Βίμπα. Ε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Αν όχι, τότε θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη και πάμε το πρώτο τμήμα στην έκθεση της κυρίας Γκόμες ε, Συμφωνία πλαίσιο εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τη Δημοσιοδημοκρατία τη Ινδονησία όσον αφορά θέματα που αφορούν την επανεισδοχή. Εδώ υπάρχουν κατ' ουσίαν δύο συμφωνίε επανεισδοχή. Ε, η πρώτη αφορά ε, την Ινδονησία και η δεύτερη συμφωνία αφορά ε, πολλές άλλες χώρες. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο πρώτα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο και κατόπιν στην εισηγήτρια την κυρία Γκόμες. Ε, καταρχήν λοιπόν να δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελα να δώσω το λόγο καλύτερα στην Προεδρία για να σας ενημερώσει τι ακριβώς συζητήθηκε στο Συμβούλιο για αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως εφόσον συμφωνείτε. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Εντάξει. Ε, το Συμβούλιο παρακαλώ, ε, σας ερωτώ, επιθυμείτε το λόγο. Αν ναι, σας τον δίνω. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο που ε, ενέκρινε αυτές τις συμφωνίες χωρίς καθυστέρηση. Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω ε, το σύνολο της συμφωνίας και να εστιάσω την προσοχή μου περισσότερο στο να σας εξηγήσω γιατί υπήρχε στο Συμβούλιο αυτή η διάσταση απόψεων. Ίσως ε, με τον τρόπο αυτό απαντηθούν ε, κάποιες ερωτήσεις του Κοινοβουλίου. Όπως ξέρετε λοιπόν οι συμφωνίες αυτές καλύπτουν μια ολόκληρη σειρά θεμάτων και ένα εξ αυτό αφορά στην επανεισδοχή. Γι' αυτό εξάλλου βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Το θέμα της ε, επανεισδοχής ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Συμβούλιο. Επειδή λοιπόν υπάρχει αυτή η ρήτρα επανεισδοχής και στις δύο συμφωνίες, θέλω να πω ότι δεν πρόκειται απλά για μια συμφωνία συνεργασίας με αυτές τις χώρες, αλλά πρόκειται για την υποχρέωση επανεισδοχής. Αυτό είναι μια νομική ρήτρα. Και χρησιμοποίησαμε βέβαια μια διαφορετική νομική βάση για να συμπεριληφθεί αυτή η ρήτρα στη συμφωνία. Εφόσον λοιπόν είναι μια διαφορετική νομική βάση, έπρεπε να ε, υιοθετήσουμε στο Συμβούλιο και μια διαφορετική διαδικασία αναγνώρισης. Ε, γιατί λοιπόν επιλέξαμε αυτό, αυτή τη συγκεκριμένη νομική βάση, αυτό όπως σας είπα έχει σχέση με την υπηρεσιδοχή. Αυτή είναι μία διαδικασία και μία άλλη διαδικασία που αφορά στην ε, υιοθέτηση των νομικών διατάξεων. Πάντως, Ακόμα και αν έχουμε αυτές τις δύο διαφορετικές ε, διαδικασίες, έχουμε μία συμφωνία. Μία συμφωνία με την Ινδονησία και μία συμφωνία με όλες τις άλλες χώρες. Και από το Συμβούλιο ζητάμε τη συνένεσή του για κάθε μία από αυτές τις συμφωνίες ξεχωριστά. Ε, πραγματικά λοιπόν ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα συνενέσει, διότι όπως ε, σας είπα αυτές οι δύο συμφωνίες κατ' ουσίαν αφορούν στη συνεργασία μας με αυτές τις δύο χώρες και βοηθούν και μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε περισσότερο ε, στο θέμα της επανεισδοχής που είναι ένα σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αν έχετε κάποιες ε, ερωτήσεις ε, προφανώς το Συμβούλιο και η νομική του υπηρεσία είναι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να συμπληρώσω και εγώ, κάτι, να εξηγήσω κάτι. Στο περιεχόμενο του άρθρου 34 που αποκόπτεται από το σύνολο της ε, υπόλοιπης ε, συμφωνίας. Όσον αφορά λοιπόν το περιεχόμενο θέλω να πω το εξής ότι εδώ μιλάμε για μια μόνιμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι γενικότερα τα θέματα της μετανάστευσης να εντάσσονται στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένας τρόπος για να γίνεται αυτό είναι να συμπεριλαμβάνονται αυτές οι διατάξεις σε ε, συμφωνίες συνεργασίας και εταιρικές σχέσεις, να υπάρχει ένα κεφάλαιο δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων. Εκεί περιλαμβάνεται ένα άρθρο μετανάστευσης και αυτό το άρθρο περιλαμβάνει τη ρήτρα επανεισδοχής. Ε, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για το άρθρο 34 παράγραφος 3. Το περιεχόμενο αυτής της διάταξης ε, είναι πολύ περιορισμένο ε, που δεν, δεν συγκρίνεται με την συμφωνία επανεισδοχής. Αυτή η ρήτρα επιτυγχάνει το εξής, επιβεβαιώνει το διεθνές, τη διεθνή νομολογία με την έννοια ότι τα κράτη πρέπει να, επαν να ε, δέχονται να, να δέχονται την επαναπρόθεση των ε, υπηκών τους. Ε, άρα δηλαδή θα πρέπει καταρχήν τα κράτη να τους εντοπίζουν τους υπηκόους του κράτους ε, και μετά να τους δέχονται χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αμελητή, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες. Αυτή κατ' ουσίαν είναι ε, και η συμφωνία. Αυτό είναι το περιεχόμενο της ε, συμφωνίας. Η κυρία Γκόμες. ήθελα να πω ότι στην υπεύθυνη για την έκθεση του Κοινοβουλίου που θα συνενέσει στην εκτενή εταιρική σχέση και συνεργασία καθώς και συμφωνία μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου. Αυτή η συμφωνία πλαίσιο ε, περιέχει το άρθρο 34 που αποτελεί τη βάση για την συμφωνία αυτή επανεισδοχής. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική η συμφωνία αυτή, διότι σε γενικούς όρους και ιδιαίτερα ως προς την επανεισδοχή, διότι είναι η πρώτη που προωθούμε με μια ασιατική χώρα και δεν είναι μια οποιαδήποτε ασιατική χώρα, είναι η μεγαλύτερη η τέταρτη πολυπληθέστερη, μια χώρα που έχει άμεση σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι ήταν μια πρώην απικία της Ολλανδίας. Και ακόμα και πριν υπήρχαν σχέσεις με τη δική μου τη χώρα, την Πορτογαλία. Είναι μια χώρα με, την, με το μεγαλύτερο ε, πληθυσμό ανά τον κόσμο για αυτή την έκθεση, 250 εκατομμύρια ε, κατοίκους. Είναι δημοκρατία πλέον και μια χώρα η οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί στις διεθνείς δεσμεύσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης είναι διαμετακομιστική χώρα για τους μετανάστες, ιδιαίτερα από, για αυτούς που προέρχονται από την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλοι ε, περνούν από την Ινδονησία για να μεταβούν στην Αυστραλία. Βεβαίως υπάρχουν ε, πολλοί όροι διότι αυτή η χώρα έχει 17.000 νησιά, υπάρχουν ε, πολλοί boat people Πολλοί βεβαίως βρίσκουν το θάνατο με την ναυσιπλοεία, γι' αυτό χρειάζονται Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να μεταβούν οι άνθρωποι από ένα μέρος του κόσμου σε ένα άλλο. Επίσης είναι μια χώρα που έχει έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, όχι μόνο λόγω γεωγραφικής θέσης αλλά και ιστορίας. Υπάρχει μια μεγάλη κινέζικη παρικία, που ζει εκεί εδώ και αιώνες. Έχουν ε, πάρει την υπηκότητα, έχουν λάβει την υπηκότητα και όταν έγινε ανεξάρτητη η Ινδονησία, πολλοί έχουν διπλή υπηκότητα, αν και αυτό δεν είναι αποδεκτό, όμως έμπρακτα αυτό συμβαίνει. είναι μια χώρα που έχει μεγάλη σημασία για τις μεταναστευτικές ροές ανά τον κόσμο όπου ε, ε, εμείς προβάλλουμε και αρρωγή για να αντιμετωπιστούν και οι παράνομοι μετανάστες και όσοι αποζητούν άσυλο. Γι' αυτό αυτή η συμφωνία επανεισδοχής έχει νόημα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 34 παράγραφος 3 της ε, συμφωνίας αυτής όπου γίνεται λόγος για επανεισδοχή. Επίσης για τους απάτριδες μπορούν, μπορεί να παρασχεθεί ε, άσυλο και για, τις, ε, για αυτούς που προέρχονται από τρίτες χώρες. Νομίζω ότι αυτή η συμφωνία θα βοηθήσει την κινητικότητα των ανθρώπων, ενώ παράλληλα έχει μεγάλη σημασία έτσι ώστε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγχει αυτές τις κινήσεις. Το Κοινοβούλιο όταν συνενέσει θα ελέγξει την εφαρμογή αυτό είναι βασικό μέλημα της, της Επιτροπής, αλλά θα συνεπικουρήσει και το Κοινοβούλιο. Έχει προωθηθεί ο διάλογος για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ Ινδονησίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει αρχίσει αυτός ο διάλογος. Θα, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό τον διάλογο σε σχέση με την ε, μετανάστευση Άρα θα ήθελα να συνενέσει το Κοινοβούλιο η Επιτροπή και το ε, Συμβούλιο θα πρέπει να μας πούν κατά πόσο περιλαμβάνονται και οι πίκοοι ε, τρίτων χωρών, ιδιαίτερα όσων κατέχουν ε, βίζα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκόμες, το Συμβούλιο και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Γκόμες για αυτή την έκθεση και για τις ερωτήσεις. Η ίδια η συμφωνία δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση επανεισδοχής υπηκών από τρίτες χώρες, αλλά στην παράγραφο 4 μιλάμε για μια ξεχωριστή συμφωνία επανεισδοχής που ήδη ενυπάρχει και θα πρέπει να υπάρχει και υποχρέωση για κατοίκους προέλευσης τρίτων χωρών. Ευχαριστώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολλά, πολύ λίγα έχω να προσθέσω. Η Προεδρία έχει απόλυτο δίκιο. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 αναφέρεται στους απάτριδες και υπηκόους τρίτων χωρών, έτσι μπορούμε στο μέλλον να ορίσουμε μία πλήρη συμφωνία επανεισδοχής, ιδιαίτερα για τους απάτριδες. Η παράγραφος 3 δεν το κάνει αυτό. Αυτό αφορά μόνο τους κατοίκους ε, τρίτων χωρών. Είναι μία ε, ρήτρα επανεισδοχής που δεν έχει καμία σχέση με τη συμφωνία επανεισδοχής που έχει 22 άρθρα. Είναι ένα, μια πολύ βασική δέσμευση που σχετίζεται μόνο για τους υπηκόους. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο όχι. Άρα το λόγο έχει η κυρία Γκόμες. Άρα, συνενώντας την Συμφωνία δοχής συμφωνούμε πρωταρχικά στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, ιδιαίτερα με τους υπηκόους και τους απάτριδες. Έτσι κατανοώ το κείμενο, έτσι δεν ερμηνεύεται. Ε, απάντηση από την Επιτροπή. Το άρθρο 34, παράγραφος 4, δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας του Συμβουλίου που έχετε ενώπιόν σας. Είναι όμως ε, μία ρήτρα δημιουργίας δυνατοτήτων, όπου τα συμβαλόμενα μέρη θα διαπραγματευτούν στο μέλλον εάν ένα από τα συμβαλόμενα μέρη το κρίνει αναγκαίο για μια πλήρη επανεισδοχή, κάτι το οποίο περιλαμβάνει τους υπηκόους τρίτων χωρών και τους απάτριδες, διότι θα είναι μια πλήρη συμφωνία. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε στο μέλλον αν χρειαστεί κάτι τέτοιο ή αν ζητηθεί. Υπάρχουν ερωτήσεις όχι. Όταν ε, γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση σε αυτή η συμφωνία θα επανέλθει στο, Κοινοβούλιο. Και με αυτή τη διασάφηση μπορώ να πω ότι ε, θα ήθελα να συνενέσουμε στο πλαίσιο αυτό, δηλαδή στα στοιχεία που εντάσσονται στη συμφωνία πλαίσιο. Ωραία. Πάμε στο επόμενο σημείο της σας διάταξης. Εδώ έχουμε η συγγήτρια τη Ρενάτα Βέμπερ είναι μία άλλη διαδικασία επανεισδοχής, δηλαδή Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών Κεντρικής Αμερικής. Η Επιτροπή ΛΥΜΠ πρέπει να εκφραστεί στο άρθρο 49 ε, σημείο 3 της διαδικασίας της Συμφωνίας Συνεργασίας για τη μετανάστευση και διαδικασία επανεισδοχής. Ε, ζητείτε η έγκριση της θέσης ε, θα πρέπει να εγκριθεί τον Ιανουάριο, έχουμε λίγο χρόνο και επειδή από την πρώτη διαβούλευση, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2003 και την ε, διαδικασία συνένεσης 10 χρόνια μετά, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ορισμένα ζητήματα. Να ζητήσουμε ορισμένες διευκρινήσεις από το Συμβούλιο, πώς εξελίχθηκε η κατάσταση καθώς και ο διαχωρισμός ως προς το τη συνεργασία 49 στο 41,3, ενώ η ΑΦΕΤ είναι υπεύθυνη για το υπόλοιπο τμήμα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο διαχωρισμός αρμοδιότητα μεταξύ ΛΥΜΠΕ και ΑΦΕΤ. Εμείς θα ασχοληθούμε ασχοληθούμε μόνο με θέματα επανεισδοχής και όχι επί των άρθρων 48 και 49. Δίνω το λόγο στην κυρία Βέμπερ καταρχήν και μετά θα ζητήσω από το Συμβούλιο να λάβει το λόγο. Καθώς και την ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Βέμπερ. Uh, thank you very much, Madam Chair. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μια συμφωνία που συζητείται από το Κοινοβούλιο, του Συμβούλιο και την Κομισιόν εδώ και δέκα χρόνια. Για να δούμε δηλαδή πόσο γρήγορα συνάπτουμε συμφωνίες. Εντάξει, είναι μια διεθνή συμφωνία και απαιτεί την ε, έγκριση των Εθνικών Κοινοβουλίων. Χρειάζεται λοιπόν κάποιος χρόνος αλλά θα ήθελα να μάθω κατά πόσον θα τεθεί σε ισχύ κατά όσο ενώ θα ζω. Ήμουν σκιώδης ηγήτρια στην ΑΦΕΤ για αυτές τις συμφωνίες και συμφώνησα με την έκθεση που συντάχθηκε για την στήριξη της ε, συμφωνίας και το γεγονός είναι ότι μιλάμε μόνο για το κομμάτι της επανεισδοχής. Μόνο τα άρθρα που αφορούν ε, επανεισδοχή και αμοιβαίες υποχρεώσεις ε, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της Κεντρικής Αμερικής. Θα ήθελα να ακούσω το Συμβούλιο και την Κομισιόν και να μιλήσω μετά για το πώς πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε <clears throat> και πώς κρίνουν ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ειδικά στο κομμάτι της επανεισδοχής και πόσο πιθανόν ή εφικτόν είναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή για το θέμα της ε, απαλλαγής των θεωρήσεων για τους υπηκόους των κρατών. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που θέσατε το ζήτημα αυτό στη μέσα διάταξη. Έχει πάρει αρκετό χρόνο για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα. Χρειάστηκε πολλής χρόνος διότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει την ανησυχία του για το θέμα αλλά το Συμβούλιο αποφάσισε να χωρίσει την διαδικασία, όπως εξήγησε και με την Ινδονησία, το ίδιο έγινε και με την παρούσα συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν το Κοινοβούλιο στο Κοινοβούλιο ζητείται για μια ακόμη να δώσει την συνένεσή του σχετικά με την συμφωνία. Αυτή ε, ο χωρισμός στα δύο τη ε, συμφωνίες ε, οφείλεται στο ότι η υποχρέωση επανεισδοχής έχει διαφορετική νομική βάση σύμφωνα με την νέα συνθήκη και Η συμφωνία αυτή επίσης περιέχει και κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν το τομέα δικαιοσύνης και ελευθερίας και γι' αυτό λοιπόν <clears throat> απαιτήθηκε αυτός ο χωρισμός των δύο ζητημάτων. Και φυσικά δεν επηρεάζει διόλου τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ούτε τις εξουσίες του σχετικά με την ε, έγκριση της συμφωνίας. Επίσης, ε, αν μου επιτρέπετε να δώσω το λόγο στην νομική υπηρεσία που ενδεχόμενα να σας διαφωνήσει περισσότερο για κάποια τεχνικά κομμάτια. Ευχαριστώ. Μερικά λόγια για να εξηγήσω αυτόν τον, ε, αυτή τη διαφοροποίηση. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να δούμε είναι ότι το Συμβούλιο κρίνει πως το ζήτημα δεν αφορά μόνο το κείμενο της συμφωνίας αλλά και το κείμενο των αποφάσεων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν επανέρχομαστε στο Κοινοβούλιο για τρίτη φορά. Κάτι ακόμα για τους λόγους αυτού του διαχωρισμού. Η συμφωνία δεν περιέχει ρήτρα περί επανεισδοχής, ούτε άλλες ρήτρες που να αφορούν τα θέματα ΔΕΗ, αλλά και ρήτρε που δεν περιέχουν κάποιες νομικές υποχρεώσεις. Πρόκειται για γενικής φύσης δεσμεύσεις, θέματα πολιτικού διαλόγου ή συνεργασίας και επειδή υπάρχει μια ρήτρα η οποία προκαλεί ε, σαφείς νομικές δεσμεύσεις τώρα θα πρέπει να αναφορωθούμε σε ε, άρθρο της συνθήκης που ονομάζεται ε, γι' αυτό ονομάζεται και νομική βάση μιλάμε για την παράγραφο 79 παράγραφο 3 που προβλέπει το δικαίωμα σύναψης συμφωνιών στον τομέα της επανεισδοχής ενένωση και 79-3 είναι τμήμα του κεφαλαίου 5.3 συνθήκε συνθήκες περί λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το σχετικό πρωτόκολλο προβλέπει ε, τη δυνατότητα για τα τρία κράτη, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, να μην λαμβάνουν μέρος σε μέτρα, είτε πρόκειται για νομοθετικές πράξεις, είτε για διεθνείς συμφωνίες. Έχουν το δικαίωμα λοιπόν να μην ε, μετέχουν σε αυτές τις αποφάσεις. Αυτό σημαίνει ότι για τη ρήτρα επανεισοδοχής είτε συμφωνία με την Ινδονησία είτε για την Κεντρική Αμερική δεν λαμβάνουν μέρος λοιπόν σε αυτές τις αποφάσεις ενώ λαμβάνουν μέρος στην απόφαση η οποία αφορά όλες τις υπόλοιπες ρήτρες της συμφωνίας. Σε κάποιες από αυτές η σύνθεση του Συμβουλίου θα είναι διαφορετική στις δύο περιπτώσεις. Γι' αυτό λοιπόν από τεχνική σκοπιάς είναι απαραίτητο να έχουμε αυτές τις δύο χωριστές αποφάσεις. Αν όμως ρίξετε μια ματιά στα εκτιμώντας και των δύο αποφάσεων, τελευταία ε, εκτιμώντας διευκρινίζουν ότι οι δύο αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν παραλλήλως, ταυτόχρονα λέει. Η στάση του Συμβουλίου είναι ότι αυτός ο διαχωρισμός ε, της απόφασης του Συμβουλίου σε δύο είναι απαραίτητη έτσι ώστε να ε, είμαστε σύμφωνοι με τα, με τα πρωτόκολλα 21 και 22. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας της εξωτερικής ε, δράσης. Θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι καταρχήν που χρειάστηκαν δέκα ολόκληρα χρόνια για να επανέλθει αυτή η τόσο σημαντική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες Κεντρικής Αμερικής. Ε, είχαν υπάρξει κάποιες ε, διαπραγματεύσεις ε, για τη Συμφωνία Σύνδεσης που και αυτές όμως χρειάζονται τη δικασία επικύρωσης. Γι' αυτό λοιπόν μετά από 10 χρόνια θα ήθελα να παρακαλέσω την εισηγήτρια και τα μέλη να περάσουν και αυτή τη συμφωνία μέσα από τη διαδικασία επικύρωσης. Ο κύριος Μπαρόζο παρακολούθησε τη συνάντηση κορφή σε ΣΥΚΑ το Σάββατο και υπήρξε και μία δήλωση των αρχηγών κρατών της Κεντρικής Αμερικής όπου εκφράζεται η έκκληση αυτή η συμφωνία επειδή σας είπα έχουν μεσολαβήσει ε, ακριβώς 10 χρόνια να προχωρήσει. Λυπούμεθα πάρα πολύ που ήταν απαραίτητο να περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα με επικυρώσεις ε, και με συζητήσεις νομικής φύσεως. Ε, θα μπορούσαμε να την είχαμε περάσει στην Κορεπέρα, αλλά και πάλι σας καλώ να την προχωρήσετε και να σας ενημερώσω ότι ο πρέσβης του Παναμά είναι ο προεδρεύων αυτής της ΣΥΚΑ, εάν θέλετε να απευθύνετε σε κάποιον για να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ακριβώς όπως και στο προηγούμενο θέμα για την Ινδονησία, πιστεύω ότι και εδώ, ε, θέλω να πω, ότι και εδώ υπάρχει μια ρήτρα επανεισδοχής που εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία συνεργασίας με λιγάκι περιεχόμενο που μοιάζει με αυτά που συζητήσαμε στη συμφωνία με την Ινδονησία. Εστιάζεται ε, στην επανεισδοχή των ε, υπηκών μιας χώρας. Ε, αυτοί θα πρέπει να μπορούν να επιστρέφουν και να γίνονται δεκτοί βεβαίως με τις απαραίτητες διαδικασίες και όσοι επιστρέφουν να έχουν τα έγγραφα ταυτοποίησης και επίσης αυτή η διαδικασία να ε, συνεπάγεται και μια αμφίδρομη υποχρέωση. Αυτή λοιπόν η διαδικασία περιλαμβάνει και μια ρήτρα εξουσιοδότησης που επιτρέπει την ε, επαναδιαπραγμάτευση ε, όλων αυτό, αυτής της ρήτρας ε, στο μέλλον για να μπορούν να περιλαμβάνονται και άτομα τρίτων, υπήκοοι τρίτων χωρών. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αν τελικά φτάσουμε μέχρι εκεί, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να διαπραγματευτεί συμφωνία επανεισδοχής με κάποια από αυτές τις χώρες, θα ακολουθηθεί η πεπατημένη και έτσι η διαδικασία επανεισδοχής θα κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να να γίνει αποδεκτή. Ε, δεν ξέρω αν κάποιος επιθυμεί το λόγο, ε, από ό,τι βλέπω όχι. Κατόπιν τούτου δίνω το λόγο στην κυρία Βέμπα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι ε, εκτιμώ ιδιαίτερα για, όλα, για τις παρεμβάσεις των συναδέλφων και θα ήθελα εκ μέρους του Κοινοβουλίου να πω ότι εμείς επιθυμούμε να στηρίξουμε τη συμπερίληψη, ε, μάλλον την, ε, την ολοκλήρωση αυτής της ε, συμφωνίας. Θέλω να σας πω ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες είναι πολλές, κατανοώ αυτά όλα ίσως να χαροποιούν τους δικηγόρους, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους συναδέλφους μας στη Λατινική Αμερική ότι αυτή η συμφωνία που ήταν αντικείμενο διαπραγματεύσεων για 10 ολόκληρα χρόνια έχει τώρα επανακατατεθεί και τώρα έχουμε μια άλλη συμφωνία σύνδεσης με τις χώρες αυτές που και αυτή ολοκληρώθηκε μετά από 5 χρόνια. Εκείνη όμως η συμφωνία αφορά μόνο το εμπόριο. Γιατί για τα πολιτικής φύσεως θέματα χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία. Και από τη στιγμή που η Συμφωνία Σύνδεσης θα έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη, τότε αυτή η συμφωνία θα ισχύει μόνο για τα στοιχεία της που θα ταυτίζονται με την Συμφωνία Σύνδεσης. Αυτά πραγματικά δημιουργούν τεράστια σύγχυση και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα θέματα να τα χειριζόμαστε διαφορετικά. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε ένας διεθνής παίκτη που ε, τον υπολογίζουν οι υπόλοιποι, πρέπει να αλλάξουμε. Έχουμε 28 μέλη, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τελικά η Ένωση είναι εκείνη που εμφανίζεται ως ε, παίκτη στο διεθνές σκηνικό. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν ε, σημαντικές αλλαγές ε, διαρθρωτικής, συνταγματικής φύσεως, ό,τι πέστε τις αλλαγές αυτές όπως θέλετε, αλλά πρέπει να λάβουν χώρα. Ευχαριστούμε την κυρία Βέμπα και τώρα Θέλω να πω ότι κλείνουμε αυτό το σημείο της ημερήσης διάταξης και πάμε στο επόμενο θέμα επειδή είναι ήδη παρούσα η συγγήτρια, γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε. Πρόκειται για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Η Βαρόνη Σάρα Λατφόρτ είναι η συγγήτρια. Ε, πρόκειται για μια έκθεση όπου αναζητώνται τρόποι για να βελτιώσουμε το ε, κείμενο νομικό πλαίσιο και θα ήθελα ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια η οποία θα σχολιάσει τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για την έκθεσή της. Και μετά ε, θα αρχίσει η συζήτηση και εφόσον επιθυμούν η Επιτροπή και το Συμβούλιο να παρέμβουν βεβαίως και θα έχουν το λόγο. Η κυρία Λάτφορντ έχει το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω αυτή την ευκαιρία να ανταποκριθώ στις τροπολογίες που υποβλήθηκαν. 150 των αριθμών, μερικές και δικές μου ε, πολλές ε, αντικατοπτρίζουν τη μεγάλη συνένεση μεταξύ σκιωδών ως προς τα προβλήματα που ανακύπτουν ως προς το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Και οφείλω να ε, τονίσω την δραστήρια συμμετοχή όλων των συναδέλφων θα ήθελα να τονίσω ορισμένους βασικούς ε, τομείς όπου θέλουμε να, βρούμε, να φτάσουμε σε συμβιβασμούς. Καταρχήν η νομοθετική δράση που χρειάζεται γιατί πρόκειται για μια έκθεση νομοθετικού περιεχομένου ίδιας πρωτοβουλίας. Γι' αυτό θα θέλαμε η Επιτροπή να προβάλλει ε, το καθεαυτό νομοθέτημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να γίνει αυτό με οριζόντια μέτρα ή με βάση το πλαίσιο που προϋφίσταται. Ε, πολλοί θέλουν κατά αυτόν τον τρόπο να αλλάξει η πρόταση πλαίσιο. Ανοίγουμε όμως το κουτί της πανδώρας έτσι και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουμε. Άρα κάθε κράτος ε, μέλος θα μπορούσε να ορίσει έναν κατάλογο προτεραιοτήτων. Και άρα θα μπορούσαμε να περάσουμε στο σύστημα αμοιβαία αναγνώρισης, να περάσουμε δηλαδή από το ένταλμα στο αμοιβαίο ε, σύστημα αναγνώρισης, δηλαδή να ολιστήσουμε σε αυτό. Στην έκθεσή μου προβάλλω ένα οριζόντιο μέτρο που προβάλλω τα θεμελιώδη δικαιώματα, την αναλογικότητα, ένα μηχανισμό διαβούλευσης και όλα τα μέσα αμοιβαία αναγνώρισης, διότι ορισμένα από τα προβλήματα του εντάλματος ε, σχετίζονται με άλλους μηχανισμούς αμοιβαία αναγνώρισης, διότι υπάρχει έλλειψη εξισορρόπησης μέσα στα πλαίσια της ε, του, της ποινική δικονομίας. Μιλήσαμε για ερευνητικά μέτρα και μέτρα δίωξης τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν για να υπάρχει ε, μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο διασυνοριακό έγκλημα και την αντιμετώπιση του αλλά ε, δεν τονίζουμε τις νομικές ρήτρες διασφάλισης πάντα. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό η τροπολογία της κυρίας Αργεντίνη από τους πράσινους είναι πολύ καλή και θα ήθελα οι σκιώδεις να τη δεχτούν. Δηλαδή να μιλήσουμε για ένα οριζόντιο μέτρο για ε, έναν οριζόντιο, μια οριζόντια αναγνώριση, αμοιβαία αναγνώριση. Διαφορετικά θα ζητήσουμε να τροποποιηθεί η ίδια η απόφαση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να ακολουθήσει την οριζόντια οδό καταρχήν, αλλά δεν αποκλείουμε την απόφαση πλαίσιο καθεαυτή. Ελπίζω οι σκιώδεις να συμφωνήσουν να δεχτούν δηλαδή αυτή την προσέγγιση. Ο δεύτερος τομέας αφορά την αναλογικότητα. Στην έκθεσή μου ζητώ ε, την έγκριση της αναλογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές θα υπολογίσουν ε, την ανάγκη ε, προβολής ενός εντάλματος, ευρωπαϊκού εντάλματος ε, σύλληψης εάν ανακύψει η ανάγκη, καθώς και άλλα ε, μέσα ή μηχανισμούς αμοιβαίας αναγνώρισης. Άρα υπάρχουν τροπολογίες με τους παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη, όπως το αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή και ιδιωτική ζωή, το κόστος δίωξης και άλλα μη παρεμβατικά μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτούς τους παράγοντες ορισμένοι θέλουν ένα, ένα διπλό έλεγχο αναλογικότητας έτσι ώστε η εκτελεστική αρχή να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί με βάση την αρχή της αναλογικότητας. Εγώ το φοβάμαι αυτό διότι πιστεύω ότι θα ανατρέψει το σύστημα. Δηλαδή θα κινηθεί πέραν του, της αμοιβαία αναγνώρισης και θα ολιστήσει προς τα πίσω. Πιστεύω επίσης ότι εάν υπάρχει ε, ένα μέσο, ένας μηχανισμός αμοιβαίας αναγνώρισης τύπου εντάλματος, τότε το κράτος μπορεί να αρνηθεί. Έχει το δικαίωμα άρνησης. Άρα το πακέτο το που προτείνω συμβιβασμού είναι το ένταλμα να συνοδεύεται από μία διαδικασία διαβούλευσης όπου οι εκτελεστικές αρχές ε, ανταλλάσσουν απόψεις σε σχέση με την αναγκαιότητα ε, λήψης ε, του μέτρου πριν εκτελεστεί και βεβαίως υπάρχει και η ασφάλεια της άρνησης με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα δηλαδή την αρχή της αναλογικότητας και την ε, ερευνητική αρχή, το ένταλμα έρευνας δηλαδή, όπως συμφωνήθηκε από το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Άρα αυτή η διατύπωση οδηγεί σε μια ισορροπία, δηλαδή ε, αναλογικότητα, διαδικασία διαβούλευσης και δικαίωμα άρνησης από την εκτελεστική αρχή. Ελπίζω οι σκιώδεις να δεχτούν αυτή τη βάση εργασίας. Ένας άλλος τομέας, στον οποίο θα ήθελα να αναφερθώ, είναι το πρόβλημα που ανακύπτει από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης δηλαδή ε, να εγκριθεί πριν από την διεξαγωγή της δίκης, πριν να είναι έτοιμη η διεξαγωγή της δίκης. Δεν θα ήθελα να προβώ σε μια διαδικασία οικοτολογίας ως προς τα στοιχεία, αλλά είναι ένα μείζον ζήτημα, διότι οδηγεί στο να κρατούνται ε, πολλοί πολίτες πριν από την διεξαγωγή της δίκης. Πολλοί μετροπολογίες ε, μιλούν για το δικαίωμα ε, άρνησης επειδή δεν είναι έτοιμη η δίκη. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα και περιορίζει το, την εμβέλεια του εντάλματος άδικα, αλλά νομίζω ότι το να είναι έτοιμη η δικάσιμος, το να είναι κοντά η δικάσιμος, έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να επιληθεί έτσι ώστε άλλα συναφή μέτρα να έχουν εξαντληθεί. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν ολόκληρο το μέσο του ε, μηχανισμού ε, αμοιβαίας αναγνώρισης, έτσι ώστε να βγει το βάρος από το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψης. Θα πρέπει να έχουμε και μεταφορά αποδεικτικών στοιχείων εκεί όπου χρειάζεται και βεβαίως ο μηχανισμός διαβούλευσης θα διασαφίσει κατά πόσο η δικάσιμος είναι έτοιμη έτσι ώστε να μην έχουμε αμοιβέ αποστολές και χρήση άλλων μέσων διερεύνησης και ο μηχανισμός διερεύνησης για να δούμε πόσο κοντά είμαστε στην διεξαγωγή της δίκης και τη δίωξη καθεαυτή. Βεβαίως τα εθνικά νομικά συστήματα διαρεύουν, αλλά νομίζω ότι Αυτό που έχει σημασία στο ένταλμα είναι στην περίπτωση της δίωξης να γίνει η μεταφορά για την ποινική δίωξη. Δηλαδή όχι να γίνει κράτηση για έξι μήνες μέχρι τέσσερα χρόνια. Δεν θέλουμε απλώς να ανακρίνουμε, θέλουμε να προβούμε σε ποινική δίωξη, να έχουμε όλα τα συναφή στοιχεία. Γι' αυτό η διαδικασία διαβούλευσης έχει μεγάλη σημασία ε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι για το πόσο κοντά ε, βρισκόμαστε στη διαδικασία δίωξης και βεβαίως η εκτελεστική αρχή αν δεν είναι έτοιμη ε, και αν δεν υπάρχει αναλογικότητα υπάρχει και ο μηχανισμός προστασίας. Δηλαδή η εκτελεστική αρχή μπορεί να αρνηθεί τη δίωξη. Τι άλλο καλύπτουν οι τροπολογίες. Μίλησα για την κράτηση πριν από τη δίκη. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να τονίσουμε. Γιατί η κράτηση μπορεί να είναι μακροχρόνια και υπό κακές συνθήκες. Κάτι το οποίο διαβρώνει την ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών και μπορεί να οδηγήσει στην άρνηση ε, δίωξης. Αυτό το πρόβλημα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε και θα ήθελα η Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την κράτηση πριν από τη διεξαγωγή δίκης, διότι ε, αυτά τα μέτρα διαβρώνουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έχω υποβάλει και εγώ τροπολογίες όπως και οι συνάδελφοι, έτσι ώστε να να ενισχύσουμε τα δίκτυα αμοιβαίας αρρωγής των συνηγόρων και να υπάρχει και να ενισχυθεί και ο, και ο μηχανισμός αμοιβαιότητας. Ελπίζω μέσα στις επόμενες ώρες να προτείνω τροπολογίες συμβιβασμού. Αύριο θα συνεδριάσουμε με τους σκιώδεις και ελπίζω να επιτελεστεί πρόοδος και οι συνάδελφοι μέχρι τότε να δουν τις τροπολογίες. Η ψηφοφορία στη ΛΥΠΕ θα γίνει τη Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. Έχουμε ορισμένα ε, σημεία που θα πρέπει να πείσω, όπου θα πρέπει να πείσω τους συναδέλφους για το πακέτο μου και την προσέγγιση μου αλλά όλων οι τροπολογίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε κυρία Λάντφορτ. Ε, Ζίπλερ και Σαρτζεντίνη θα λάβουν το λόγο σκιώδης και επειδή και εγώ είμαι σκιώδης θα ήθελα να πω πολύ λίγα λόγια. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω, όπως αναφέρθηκε επανειλημμένα, ότι ένα από τα σημαντικότερα νομικά εργαλεία που ισχύουν στον τομέα της ε, δικαστικής ε, συνεργασίας είναι αυτό ακριβώς το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Δικαστική λοιπόν συνεργασία σε ποινική φύσεως ε, θέματα και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Όπως είπε και η κυρία Λάτφορτ, θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό, ότι εδώ ε, πρόκειται ή το ένταλμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται οποτεδήποτε πρόκειται για ποινικά αδικήματα και θα βασίζεται στην αρχή της αμοιβαία ε, αναγνώρισης. Γιατί είναι ένα εργαλείο αμοιβαία αναγνώρισης. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι δεν πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο αυτή την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Ακούγοντας αυτά που είπατε, άκουσα ότι συμφωνείτε κι εσείς ε, μαζί μου. Στηρίζω ανεπιφύλακτα την προσέγγιση της εισηγήτριας ε, σε όλα σχεδόν τα σημεία που έπτυξε. Επίσης ε, συμφωνώ ε, σε αυτό που είπε ότι ανησυχεί μήπως ανοίξει το κουτί της Πανδώρας και σε αυτό συμφωνώ ε, και στο θέμα του ελέγχου της αναλογικότητας και επίσης και στο πώς θα δείξουμε το θέμα της προφυλάκησης. Θέλω λοιπόν ε, να επισημάνω ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί για συμβιβασμούς, ε, στηρίζω ανεπιφύλακτα την προσέγγιση της εισηγήτριας σε όλα αυτά τα θέματα. Βεβαίως και θα υπάρξουν ε, κάποιες τροπολογίες που δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σε γενικές όμως γραμμές θεωρώ ότι θα βρούμε τη βέλτιστη δυνατή λύση και θα μπορέσουμε να στηρίξουμε την εισηγήτρια. Η κυρία Σίπχολ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που μας έδωσε έτσι μια γενική εικόνα για όλες αυτές τις λεπτομέρειες που συζητάμε. Και εμείς θα καταθέσουμε τροπολογίες για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Βέβαια δεν θα σχολιάσω όλες τις λεπτομέρειες γιατί σε ορισμένα θέματα έχουμε την ίδια άποψη, ε, σε άλλα πάλι διαφοροποιούμεθα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα είτε με οριζόντιες λύσεις είτε ανοίγοντας το ίδιο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Το θέμα είναι το εξής. Οι πολίτες περιμένουν ξεκάθαρους κανόνες και εδώ ε, το θέμα είναι ότι έχουμε ένα ευρωπαϊκό μέσο, ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης στην ε, πράξη πρέπει να δούμε ποια είναι η κατάσταση γιατί το θέμα είναι ότι πρέπει να βασιζόμαστε στην ε, αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Υπάρχουν όμως ε, και εθνικοί κανόνες. Αυτό λοιπόν οδηγεί σε σύγχυση όχι μόνο στον τομέα των ε, επαγγελματιών ε, και των θεσμών ή και στο θέμα των πολιτών. Γιατί ανεξάρτητα με το ποια είναι η κατάσταση ενός πολίτη, εάν αυτή είναι είτε είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έχουν κάποιες επιφυλάξεις. Οι πολίτες, όταν μιλάμε για ευρωπαϊκά μέτρα, οι πολίτες ε, επιθυμούν να υπάρχουν κοινά πρότυπα εναρμονισμένα και αυτά δεν υπάρχουν. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη, αυτό είναι το βασικότερο θέμα σε όλες αυτές τις συζητήσεις ε, που κάνουμε και αυτό ε, έχει και άμεση σχέση με την αποδοχή της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μέσο που σκοπεύει στο να βελτιώσει τη συνεργασία στον δικαστικό τομέα, στον τομέα ποινικών διώξεων. Απ' την άλλη όμως έχει και άμεση σχέση με τα ε, ατομικά δικαιώματα, το δικαίωμα της άμυνας, της υπεράσπισης μάλλον, ε, Άρα δηλαδή όλες οι λεπτομέρειες που συζητάμε πρέπει να δούμε κατά πόσον θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με την α ή τη β μέθοδο έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να καταλήξουμε σε κοινά πρότυπα. Όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν μιλάμε μόνο για ε, τα μέτρα και σταθμά για την δίωξη αλλά και για την υπεράσπιση που πρέπει να είναι στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο ισχύει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα να το δούμε πολύ προσεκτικά διότι αλλιώ οι πολίτες δεν θα δεχθούν ευρωπαϊκά πρότυπα ανεξάρτητα με το σε ποιο, για ποιον το μιλάμε, εφόσον τα πρότυπα αυτά βασίζονται μόνο σε εθνικούς κανόνες. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να δείξω δύο θέματα. Τον ε, έλεγχο αναλογικότητας στη χώρα η οποία καλείται να παραδώσει τον ύποπτο και δεύτερον την ανάγκη για νομοθετική πρόταση. Ξεκινάμε με τον έλεγχο αναλογικότητας. Θα σας αναφέρω συγκεκριμένο παράδειγμα γιατί κατά την άποψή μου ο έλεγχος σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αρκεί. Ας πούμε έχουμε έναν Ολλανδό που είναι στην ε, Άμστερνταμ, καπνίζει καφέ και καπνίζει, πίνει καφέ και καπνίζει και μαριχουάνα που επιτρέπεται στο Άμστερνταμ. Έρχεται ένα Σουηδός και το ρωτάει πού το βρήκε αυτό το τσιγαριλίκι και ο Ολλανδός του λέει εκεί πιο πέρα ε, σε έναν δρόμο μπορείς να αγοράσεις ε, το χασίς. Πάει ο Σουηδός, το αγοράζει, έρχεται πίσω στο καφενείο, κάθεται εκεί στο μπαλκόνι μαζί με τον ε, Ολλανδό ε, και ανάβει και αυτό το τσιγάρο του. Συζητάνε και αλλάζουν, ανταλλάσσουν και διευθύνσεις. Μετά, ε, Ολλανδός ε, πάει στη Στοχόλμα, αυτό τον κάλεσε ο άλλος, ε, δεν τα πετάει όλα αυτά που αγόρασε στο ε, Άμστερνταμ και τον συλλαμβάνουν στη Στοχόλμη γιατί φαίνει μαζί του χασίς. Ε, πανικοβάλλεται, δίνει τη διεύθυνση του Σουηδού που δεν του πούλησε όμως αυτός, απλά γνωρίστηκαν στο καφενείο και ο ε, Ολλανδός κατηγορείται ο Σουηδός εννοεί μάλλον η γεωμιλήτρια, ο Σουηδός λοιπόν ε, παίρνει και αυτό ένταλμα σύλληψης γιατί υποτίθεται ότι πούλησε. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ πρέπει να έχουμε τεστ αναλογικότητας. Η Σουηδία έχει πολύ ωραίες φυλακές, κανένα πρόβλημα, ε, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπάρχει όμως το θέμα της αναλογικότητας. Σας ανέφερα λοιπόν αυτό το παράδειγμα γιατί θεωρώ ότι ε, το τεστ αναλογικότητας πρέπει να γίνεται και στις δύο πλευρέ. Τελικά γιατί δεν πάει αυτό στη Σουηδία ο Ολλανδός γιατί δεν ήταν Ολλανδός, ήταν Σύριος τελικά που κρατείτο για πάρα πολλά χρόνια ε, σε φυλακές στη Συρία και αν τον ξανακρατούσαν ε, θα αυτοκτονούσε. Όσον αφορά τώρα την νομοθετική πρόταση, νομίζω ότι πρέπει να καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα καθιστά σαφές ότι είτε θα αλλάξουμε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή θα αναζητήσουμε οριζόντια μέτρα ε, που θα φύγουν το θέμα αλλά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και θέλω να είναι σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει μια νομοθετική πρόταση είτε μόνο γι' αυτό είτε οριζόντια ρυθμίση. Αλλά η λύση να είναι μέσα σε ένα χρόνο. Γιατί δεν μπορούμε ε, να βάλουμε έτσι μια ε, συγκεκριμένη ημερομηνία, ε, να το δούμε το θέμα στη διάρκεια ενός έτους και τότε θα δούμε κατά πόσον η έκθεση της Σάρας πράγματι επέφερε την αλλαγή που επιθυμούμε. Ο κύριος Ντεγιόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, εισηγητές και την εισηγήτρια για τη συζήτηση γιατί προκύπτουν κάποια σημαντικά θέματα. Η ε, κυρία, η κυρία έθεσε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων λέγοντας ότι ακόμα δεν υπάρχει εναρμόνιση. Δεν υπάρχει εναρμόνιση θεμελιωδών δικαιωμάτων, κυρίως ε, κατά την εφαρμογή της ποινική διαδικασίας. Εχθές είχαμε εδώ την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ η οποία μίλησε για το δικαίωμα νομικής ε, αρρωγής με την έννοια ότι έτσι τίθεται επιτάπητος και το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Αλλά δεν έχει ακόμα εγκριθεί η νομική αρρωγή και κανείς δεν περιμένει ότι ε, θα γίνει δεκτό αυτό το θέμα σε αυτή την θητεία. Επίσης να πω ότι οι συζητήσεις που είχαμε χθε με την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ σχετικά με την προτινόμενη νομοθεσία στη Ρουμανία σχετικά με την ε, διαφθορά όπου πλέον ε, η πολιτική διαφθορά δεν είναι ποινικό αδίκημα για να δούμε τι θα γίνει στην πράξη αν έχουμε ας πούμε μια διεφθαρμένη αρχή, έναν διεφθαρμένο φορέα σε ένα ε, κράτος μέλος και ζητείτε το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προφανώς και θα πρέπει να είμαστε ευτυχείς γιατί υπάρχει το θέμα της αμοιβαία αναγνώρισης. Όμως στην πράξη αυτό δεν είναι αλήθεια. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές δυσκολίες στα κράτη-μέλη και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ώστε να λέμε ότι ισχύει η αρχή της αμοιβαία αναγνώρισης και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κατά τα άλλα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι τροπολογίε μου είναι περίπου ίδιες όπως και αυτέ των πρασίνων μόνο που δεν είμαι ακόμα πεπισμένος ότι μια οριζόντια ρύθμιση ε, θα ήταν αποτελεσματική. Πρέπει να με πείσετε επ' αυτού. Θεωρώ ότι προς το παρόν τουλάχιστον πρέπει να παραμείνουμε σε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε ένα χρόνο να καταθέσει προτάσεις για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Και αν τελικά ε, χρειαστεί να τροποποιηθεί ε, το ίδιο το ένταλμα, αυτό μπορεί να είναι στη διακριτική ευχαίρεια της Επιτροπής. Όμως το μήνυμά μας πρέπει να είναι σαφές. Και ε, αύριο στις συνεδρίες των ε, σκιωδών θα συζητήσουμε για τις τροπολογίες μου. Η κυρία Ρομέρο Λόπες. Ευχαριστώ. Ήθελα να μιλήσω πάνω κάτω όπως και ο κύριος Γιόγκ, διότι εκτιμώ ιδιαίτερα την εργασία που έκανε η Σάρα Λατφόρντ, αλλά νομίζω ότι δεν θα επαρκέσει, διότι όλα τα ζητήματα της αναλογικότητας είναι αρκετά αδύναμε, αδύναμα. Υπάρχουν κράτη που δεν θεωρούν ως ε, αδίκημα κάποιες περιστάσεις που άλλα κράτη θα θεωρούν ως αδίκημα και αυτός ο κατάλογος των σοβαρών εγκλημάτων, σοβαρών δεκιμάτων που αναφέρονται στην οδηγία πλαίσιο, απόφαση πλαίσιο συγγνώμη, ε, ε, δεν ε, είναι αρκετά συγκεκριμένα και διευκρινισμένα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω κύριε Λοφόρτ ότι πολλά στην έκθεσή σας είναι επαρκή αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε μάλλον σε ένα χρόνο μια αξιολόγηση εξαντλητική ανάλογα με το τι ε, εντάλματα θα εκδοθούν κλπ. Διότι πράγματι βασιζόμαστε σε σοβαρά εγκλήματα, αλλά η ασάφεια θα έλεγα είναι κατά το μάλλον ήταν ευρεία και δυστυχώς ε, θεωρώ πως ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει κάποια μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας πλαίσιος ε, στο μέλλον διότι δεν πρόκειται να επαρκέσουν για την επίλυση του προβλήματος. Θα πρέπει να γνωρίζουμε μέσα σε ένα έτος ποια θα είναι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή αυτών των συστάσεων και αν επαρκούν. Διότι κατά την άποψή μου δεν θα είναι επαρκή, επαρκή αυτές τις συστάσεις διότι δεν υπάρχουν ε, παντού ισότιμα αδικήματα σε ό,τι αφορά την καταδίκη που επιβάλλεται, διότι η ε, τριετία δεν είναι επαρκής, θα πρέπει να είμαστε πιο σαφείς προκειμένου να μην βρεθούμε ενώπιον καταστάσεων δυσάρεστων. Εντάξει, πρόκειται ένα βήμα, ε, αλλά Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία χάρη στην εργασία της κυρίας Λάτφορτ θα ε, μπορέσουν ε, να ρυθμιστούν, αλλά δεν επαρκούν. Θα πρέπει να προβούμε σε μια μεταρρύθμιση αυτής της οδηγίας της απόφασης πλαίσιο για να περιληφθούν πιο συγκεκριμένα στοιχεία για μια έκδοση παραδείγματος χάρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στρέφουμε προς την Κομισιόν, αν θέλει να λάβει το λόγο. Η Κομισιόν είναι αρνητικά. Εντάξει, τότε ο λόγος στην κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ. Θα ήταν καλό να ακούσουμε την Επιτροπή. Χθες ε, δεν άκουσα τι είπε η κυρία Ρέντινγκ αν έχει κάποια άποψη, αν η Κομισιόν θα είναι έτοιμη να προτείνει οριζόντια μέτρα. Εν δεν ε, άκουσα κάποια απάντηση σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σίγουρα δεν μπορούσε να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που τέθηκε, αλλά θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας απαντήσει. Υπάρχει ε, συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στην Κομισιόν και το Κοινοβούλιο που διέπει τις ε, προϋποθέσεις για την απαντήσεις που πρέπει να δίνονται στις ε, πρωτοβουλίες, ε, σε εκθέσεις πρωτοβουλίες μάλλον και υπάρχει έκθεση της Αργεντίνη που ζητάει ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προσαρμοστεί μέσα σε ένα χρόνο μετά από την πρόταση αυτή. Συμφωνώ λοιπόν με την ε, ανάγκη να τεθεί κάποιο χρονικό όριο. Εάν η έκθεση περάσει, που ελπίζω πως θα περάσει, και ελπίζω να βρίσκομαι και στο επόμενο κοινοβούλιο, αυτό είναι κάτι το οποίο θα υποχρεώσει την Κομισιόν και θα να έρθει να ανταποκριθεί εντός ενός έτους. Φυσικά θα το λάβουμε υπόψη μας αυτό στις ακροάσεις ε, του Επιτρόπου για τα, για τα θέματα τα δικαστικά. Θέλουμε λοιπόν σαφείς απαντήσεις από πλευράς Κομισιόν. Ο προβολές λοιπόν θα είναι στραμμένος ε, προς την πλευρά της Κομισιόν εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να ασκήσουμε τώρα αλλά και στο εγγύς μέλλον πίεση προς την Κομισιόν. Το πρόβλημα είναι επίγον και σοβαρό. Θα πρέπει λοιπόν η διαδικασία να συνεχίσει την διαδρομή της, να μην εκτροχιαστεί. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, τακτικές για να πετύχουμε το αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουν διάφορες δυνάμεις ε, που προφανώς είναι κατά το θέμα του ευρωπαϊκού εντάλματος Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε θέση να αποδείξουμε ότι αυτές είναι εσφαλμένες θέσεις Κάποια τα προβλήματα τα έθιξαν ήδη οι συνάδελφοι. Αναφέρθηκαν προβλήματα τα οποία είναι σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση. Κοιτάξτε, η συζήτηση συνεχίζεται. Θα πρέπει να επιτευχθεί επιτυχία ανάμεσα στον παθμό εναρμόνισης που είναι διαφορετικό ζήτημα με την ε, ομοιομορφία, χρειάζεται ως εκ τούτου να έχουμε τους εθνικούς ποινικούς κώδικες οι οποίοι να είναι ισοδύναμοι, ισότιμοι κατά κάποιο τρόπο. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι επιθυμητό αλλά και δεν είναι και εφικτό. Θα πρέπει τα συστήματα να είναι ε, διαδραστικά, διαλειτουργικά και γι' αυτό τονίσαμε τόσο πολύ το ζήτημα όπως και η κυρία Σίπελ το ανέφερα. Εγώ ήμουν εισηγήτρια σε ένα, μία από τις τρεις εκθέσεις όπως η κυρία Αντωνέσκου ήταν στο τρίτο Πάντως ε, πρόοδος ε, επιτέλους ε, επιτεύχθηκε και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αλλά και να το στηρίξουμε. Τώρα η κυρία Σαρτζεντίνη ανέφερε την θέση της και μας έδωσε για ένα παράδειγμα για την ανάγκη αναλογικότητας καρδιά για τις εκτέλεσεις Νομίζω όμως ε, ότι το παράδειγμα που ανέφερε ξεπέρνει κατά πολύ την αρχή της έμβαιας αναγνώρισης. Ε, πιστεύω πως ε, ενδεχομένως όσο προχωράμε προς περισσότερα μέτρα τότε θα πρέπει να δεν τα, τις διάφορες αρχές ε, οι οποίες ε, εμπεριέχονται στις ε, αρχές των θεμελιδών δικαιωμάτων. Ελπίζω λοιπόν να τύχω της στήριξης των συναδέλφων σε αυτό το τριμερές, τριπλό πακέτο που προανέφερα και το κράτος μέλος θα πρέπει να ε, ενημερώνει για τον τρόπο εκτέλεσης ε, του εντάλματος και αν ε, τις απαιτήσεις δεν είναι ικανοποιητικές ότι οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν τα μέτρα. Αναφέρονται στο Βασίλειο, από το 2003 έχουμε νομοθετήσει. Όταν ε, πρωτεφαρμόστηκε το ένταλμα σύλληψης και αποφασίσαμε ο δικαστής να έχει την δυνατότητα να απορρίψει την εφαρμογή του. Αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερος και ένας από τους λόγους ο οποίος ε, τίθεται στο κέντρο αυτής της έκθεσης είναι να ενθαρρύνουμε τους εθνικούς δικαστές εάν όλες οι άλλες επιλογές έχουν εξαντληθεί αυτή θα είναι η τελευταία προσφυγή, η τελευταία δυνατότητα που παρέχεται στον δικαστή. Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν μια αναγνώριση εκεί να υπάρχει ως εγγύηση. Με ικανοποιεί εδώ ότι δέχεστε και συμφωνείτε σχεδόν με όλα όσα δήλωσα στην αρχική μου παρουσίαση. αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε για την διατύπωση και θα φροντίσω πριν από το γεύμα να σας υποβάλω τις προτάσεις μας και θα ήμουν ευτυχής να μπορέσουν οι συμβαστικές προτάσεις που θα κάνω να μας βρίσκουν, να μας σύμφωνος και να περάσουμε ήπια στην ψηφοφορία τον Ιανουάριο. Γνωρίζω όμως πως υπάρχουν κάποια σημεία για τα οποία δεν ε, θα έχω μπορέσει να πείσω τους συναδέλφους, αλλά φαντάζομαι πως αντίγω τη στήριξη της Ευχαριστούμε κυρία Βάντφορτ. Θα ψηφίσουμε 13 Ιανουαρίου. Θα είναι έκτακτη η συνεδρίασή μας στο Στρασβούργο και νομίζω ότι οι σκιώδεις αύριο θα έχουν ε, την ε, δυνατότητα να φτάσουν σε ένα πολύ καλό συμβασμό. Σας ευχαριστώ όλους για τη συνεργασία. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, διότι η ψηφοφορία προβλέπεται για τις 11 παρατέταρτο. Διακόπτουμε λοιπόν, γιατί πρέπει να περιμένουμε τους συναδέλφους που θέλουν ε, να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στις 10.45. Hello everybody. Γεια σας και πάλι. Ας συνεχίσουμε παρακαλώ. Συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Η πρώτη κατά της ε, παραχάραξη, έκθεση κατά της παραχάραξη. Κυρία Μάκιντάιρ δεν θέλει να λάβει το λόγο. Όχι, απλώς για να πω ότι ήταν εξαιρετική η συνεργασία με όλους τους ε, σκιώδους, σας ευχαριστώ και ελπίζω να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα έτσι ώστε να προωθηθεί ο τριμερής ε, διάλογος του χρόνου. Ωραία. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 35 αποσύρεται. 36 υπέρ. Κατά. Πρέπει να ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 36. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Πέρας. 28 υπέρ, 16 κατά, άρα εγκρίνεται. Συμβασμός 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ, κατά. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν σηκώνεται χέρι, χέρια. 38. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ 3 κατά, αλλά σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας, διαφορετικά θα πρέπει να ελέγχουμε. 39 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 40 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Σύμβασμος 5 υπέρ κατά. Πρέπει να ελέγξω. Συμβάσμος 5. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 27 υπέρ, 19 κατά, καμία αποχή, άρα εγκρίνεται. Έκον 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, υπέρ, πάλι παρακαλώ, κατά, αποχές Εγκρίνεται με πλειοψηφία. 44 υπέρ. Α, είναι πανομοιότυπη, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε. 44 και 45. Τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 46 υπέρ. Α, όχι, καταπίπτει. Συμβασμός 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 55 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 12 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 13 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 14 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία υπέρ, ε, τα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά πρέπει να ελέγξουμε την 12 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας 24 υπέρ 23 κατά άρα εγκρίνεται Δεν αλλάζει η έκβαση της ψηφοφορίας, ακόμα και με τη δική σας ψήφο. Έκον 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έκον 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. 15. Ωραία, ελέγχουμε. Ελέγχουμε γιατί 14. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 25 υπέρ, 22 κατά, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 1 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έκον 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 και 21 είναι πανομοιότητες υπέρ. Α, 20 καταπίπτην, ναι, έχετε δίκιο. Άρα, συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έκον 4 κατά τι άρα 32 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συνδυασμός 4 που καλύπτει την 1 και 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και μετά ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί. Θα ήθελα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 46 υπέρ κανείς κατά, δύο αποχές και τώρα θα πρέπει να ψηφίσουμε, να αρχίσουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αρχίζει ε, η ψηφοφορία, χρειαζόμαστε 31 ψήφους υπέρ. Πέρας. Είναι σαφές 46 ε, υπέρ ουδής κατά δύο αποχές. Κυρία Μακιντάιερ, συγχαρητήρια. Τώρα στρεφόμαστε στην έκθεση ε, για τον γενετήσιο προσανατολισμό. Κυρία Λούνατσεκ, θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ εντάχει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης για την ε, πολύ επικοδομητική συνεργασία. Ξέρουμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά είχαμε πολύ καλούς συμβιβασμούς και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις της ομάδας, όλων των ομάδων που υποστήριξαν την έκθεση αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ και στο κείμενο που προέρχεται από την Επιτροπή ΦΑΜ Εκεί είδαμε ότι οι περισσότερες ε, τροπολογίες που υπερψήφισε η Επιτροπή καλύπτονται από το δικό μας κείμενο. Υπήρχαν δύο που θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο κείμενο που έχετε στον κατάλογο ψηφοφορίων. Ελπίζω να τα καταφέρουμε πολύ καλά και εδώ και στην Ολομέλεια αργότερα. Ευχαριστούμε κυρία Λούνατσεκ. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά.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 κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Υπόδειξη 7 υπέρ. Α, με συγχωρείτε. 14, 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται.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 Υπόδειξη 8. Υπέρ. Άλλη μια φορά. Γιατί δεν ψηφίζεται. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Υπόδειξη 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Θέλετε να ελέγξουμε, ελέγχουμε την 25. Αρχίζει η ψηφοφορία. 25. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 31 υπέρ, 13 κατά, 3 αποχές, άρα εγκρίνεται. Τροπολογία. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Υπόδειξη 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να ελέγξουμε. Υπόδειξη 4. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 24 υπέρ, 22 κατά, μία απόδειξη, άρα εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, 30 με συγχωρείτε υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Υπόδειξη 15 υπέρ, κατά,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 Καμία αποχή, άρα απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός τροπολογίας 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Υπόδειξη α υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Υπόδειξη β Α, καταπίπτει, ωραία. Άρα ψηφίζουμε το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. 40 υπέρ, κατά 2 και 6 εποχές. Άρα εγκρίνεται και συγχαρητήρια στην κυρία Λούνατσεκ. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, η τελευταία μας ψηφοφορία, για τη δέσμευση και δίμευση προϊόντων του εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Μάκοβα, θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εντάχει, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις ιδιαίτερα για τη σκληρή εργασία και τις πολύ καλές συμβουλές και θα ήθελα να πω ότι η Λιθουανική Προεδρία μας βοήθησε ιδιαίτερα και πίεσε το Συμβούλιο να, να τελειώσει, να ολοκληρώσει τον τριμερή διάλογο. Εγώ δεν έφτασα στους στόχους, όλους τους στόχους που επιθυμούσα, αλλά έγιναν βήματα προς τα εμπρός και έχουμε ενώπιόν μας το κείμενο το οποίο βρίσκει όλους σύμφωνους. Τελική ψηφοφορία για το ε, κείμενο. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία για ολόκληρο το κείμενο. Πέρας. 44 υπέρ, ένας κατά μία αποχή. Να συγχαρούμε την κυρία Μακοβέ. And this was for, for today's vote. Αυτά για σήμερα. Επειδή όλα τα άλλα σημεία αναβλήθηκαν, θα συνεχίσουμε στις 3 το απόγευμα, στις 3 με, την, με τον απολογισμό της Λιθουανικής Προεδρίας. Σας ευχαριστώ συνάδελφοι.